Αγαπητοί συνάδελφοι, θα συνεχίσουμε. Καταρχήν θα ήθελα να σας δείξω συγγνώμη γιατί σήμερα το πρωί δεν ε, τηρήσαμε ενός λεπτού συγγύη για τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων στο Λονδίνο. Παρακαλώ να με συγχωρέσετε που σήμερα το πρωί δεν τιμήσαμε τα θύματα. Ίσως θα ήταν καλό να μας το έχει επισημάνει στην αρχή της συνεδρίασης και θα το κάναμε. Δεν ήταν κακή πρόθεση από μας, αλλά εάν αυτό επαναληφθεί, παρακαλώ να μας το επισημάνετε εν συντομία. Και τώρα θα περάσουμε στο σημείο 12, την ανταλλαγή απόψε με το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που καλωσορίζω την κυρία Ιβάνοβα εδώ. Το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο τους προηγούμενους μήνες ε, εκπώνησε μια σειρά από δικές εκθέσεις, ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης και ειδικά μέτρα απασχόλησης για τους νέους, τόσο στον τομέα της ε, ανεργίας των νέων. Ε, και χαίρομαι πολύ που η κυρία Ιβάνοβα βρίσκεται εδώ για να μας πει κάποια πράγματα για τα αποτελέσματα του, της εργασίας στο ελεγκτικό συνέδριο. Νομίζω ότι μπορεί όλα αυτά να είναι πολύ χρήσιμα για την δική μας εργασία και θα μπορέσουμε να τα συμπεριλάβουμε στις δικές μας προτάσεις ούτως ώστε να χρησιμοποιήσουμε πιο αποτελεσματικά τους ισχνούς πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας. Νομίζω ότι οι επισημάνσεις μας είναι εξαιρετικά, οι σας είναι εξαιρετικά χρήσιμες για μας. Γι' αυτό σας δίνω το λόγο θα έλεγα για ένα τέταρτο, ούτω ώστε να μείνει λίγος χρόνος μετά ε, για τη συζήτηση. Έχετε το λόγο, κυρία Ιβάνοβα. Είναι μεγάλη χαρά, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, να είμαι ε, εδώ για πρώτη φορά το ελεγκτικό συνέδριο έχει προσκληθεί στην Επιτροπή Πολιτισμού. Είναι πολύ μεγάλη χαρά να σας παρουσιάζουμε κάποια από, τα, τις ειδικές μας εκθέσεις ε, που ε, για την οποία είμαστε διάσημοι αυτή η ειδική έκθεση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, αλλά αφιερώνουμε και πολύ χρόνο, προσπάθεια και έργο στην ειδική μας έκθεση που ασχολείται με τις επιδόσεις. Αυτό που είπατε ακριβώ, κυρία Πρόεδρε, η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα της οικονομίας, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που, που έχουν ε, προκύψει από ε, τα ευρωπαϊκά ταμεία, ε, και επειδή είμαι και πρώην μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι μεγάλη χαρά για μένα να ε, παρίσταμε σήμερα στην Επιτροπή ε, Πολιτισμού είναι μικρή η οικονομική ανάκαμψη και αυτό ακόμη περισσότερο δείχνει πόσο σημαντική είναι ε, οι ε, πόσο σημαντική είναι η ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών. Για ποιο λόγο είναι η εκπαίδευση σημαντική, ειδικότερα για αυτήν την Επιτροπή, δεν χρειάζεται να το εξηγήσω. Ε, κανείς δεν μπορεί να τονίσει αρκετά τη σημασία της εκπαίδευσης, ε, το βλέπουμε αυτό, το επίπεδο της εκπαίδευσης έχει άμεση σχέση με την απασχολησιμότητα. Κατά τα πρόσφατα έτη η απασχόληση ήταν ε, τρεις φορές μικρότερη ε, για, για, εκείνους που είχαν ανώτερη εκπαίδευση σε με αυτούς που είχαν ε, πρωτοβάθμια εκπαίδευση μόνο. Νομίζω ότι η εκπαίδευση έχει πολύ μεγάλη σημασία για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη καθενός ε, και έχει άμεση σχέση και με την ποιότητα της ζωής. Άλλα ωφέλη όπως ε, Καλύτερη συμμετοχή ε, του πολίτη στα κοινά και βελτιωμένες συνθήκες υγείας είναι επίσης πολύ σημαντικές. Μπορούμε να περάσουμε στις επόμενες διαφάνειες. Ε, είναι πάρα πολύ βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης η προώθηση της εκπαίδευσης και η βελτίωση της πρόσβασης σε αυτή. Ε, στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να ενισχύσει τα κράτη-μέλη και να τα συντονίσει που έχουν μία πλήρη αρμοδιότητα και αποκλειστική για τις εκπαιδευτικές πολιτικές. Όπως βλέπετε από την ε, ε, γραφική παράσταση, ε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, η εθνική συνεισφορά στην εκπαίδευση μεταξύ 2007 και του 2011 ήταν περίπου 3,2 δις και η ε, ε, συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι περιορισμένη, όμως είναι σημαντική σε απόλυτους όρους. Βλέπετε 33,7 δις για την περίοδο 2007 με 2013 και βλέπετε από το 2014 μέχρι το 2020 είναι γύρω στα 27,1 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Επειδή η εκπαίδευση είναι πολύ ευρύ θέμα, ε, για το δικό μας έλεγχο επικεντρωθήκαμε ε, στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που ήθελε να επιτύχει η συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Είναι η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αύξηση της συμμετοχής της διαβίου μάθησης, μείωση του αριθμού όσων έχουν χαμηλές επιδόσεις, βασικές δεξιότητες, ε, εμείς καλύψαμε περισσότερο τους στόχους που αφορούν την εκπαίδευση και την κατάρτιση για το πλαίσιο του 2010 και του 2020, όπως επίσης και στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ευρώπη, για τη στρατηγική για το 2020. Βλέπουμε ποια ήταν τα κριτήρια που ε, χρησιμοποιήθηκαν για να μπορέσουν να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, κατά πόσο οι στόχοι επετεύχθησαν ε, στα επιχειρησιακά προγράμματα μέχρι το 2020, όπως επίσης ε, κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστήριξε τα κράτη-μέλη ε, κατά ε, την, ε, τον καθορισμό του τρέχοντος προγράμματος, θα μας πάει μέχρι το 2020, στο πλαίσιο δηλαδή του επιχειρησιακού προγράμματος, με σκοπό να το βελτιώσουμε και κάνουμε και σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο. Στον έλεγχό μας λοιπόν είδαμε 37 επιχειρησιακά προγράμματα για την περίοδο 2007 μέχρι 2013 από 17 κρατημέλη, περίπου 83% του συνολικού προγράμματος ε, υποστήριξης εκπαίδευση από το 2007 ω το 2013. Ε, είδαμε επίσης και πέντε συμφωνίες εταιρική σχέσης ε, του τρέχοντος προγράμματος και η αξιολόγησή μας επικεντρώθηκε σε πέντε κράτη-μέλη, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ρουμανία. Τα περισσότερα κονδύλια δαπανήθηκαν σε αυτές τις χώρες και είδαμε και κάποια άλλα κριτήρια γεωγραφικής ισορροπίας κλπ. Ε, τρεις ε, προγράμ, τρία, προγράμματα από το, τρία προγράμματα από το προηγούμενο, την προηγούμενη προγραμματική περίοδο εξετάσαμε. Ε, θεωρήθηκαν βέλτιστες πρακτικές ε, κατόπιν συστάσεων των κρατών μελών. Εμείς Στην επόμενη διαφάνεια βλέπουμε την αξιολόγηση ε, του των προγραμμάτων επιχειρησιακών από το 7 ως το 13. Η ανάλυση μας ε, του επιχειρησιακού αυτού προγράμματος ε, έδειξε ότι σε γενικές γραμμές οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ελήφθησαν υπόψη και συμπεριλήφθηκαν. Βέβαια, Κάποια στοιχεία των, ε, της λογικής παρέμβασης ε, δεν αναπτύχθηκαν επαρκώς. Ποια είναι η λογική παρέμβαση. Ε, τα επιχειρησιακά προγράμματα είναι στρατηγικά έγγραφα που στηρίζουν την παρέμβαση της Ένωσης, αλλά δεν περιλαμβάνουν διεξοδική πληροφόρηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμω πρέπει να αξιολογήσει και να τα βελτιώσει, δηλαδή να δοθεί απαραίτητη πληροφόρηση σε σχέση με τη λογική πίσω από αυτήν την παρέμβαση της Ένωσης. Αυτή είναι η βάση λοιπόν για την ε, χορήγηση των ε, ε, κονδυλίων Όσον αφορά την περίοδο από το 2007 έως το 2013, το ελεγκτικό συνέδριο αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα στοιχεία. Είπε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν σε δύσκολη θέση για την αποτελεσματική και επαρκή παρακολούθηση της ε, συνολικής επίδοσης λόγω του ρυθμιστικού ε, προγράμματος. Ε, ήταν απαραίτητο να δει κανείς τον αριθμό των συμμετεχόντων, αλλά δεν υπήρχαν κοινοί δείκτες, κάτι το οποίο βέβαια δεν επιτρέπει την ομοδοποίηση των ε, αποτελεσμάτων παρακολούθησης. Όσον αφορά τώρα την περίοδο ε, που αφορά τη στρατηγική για την Ευρώπη το 2020 ε, είχε λίγο αντίκτυπο ως προς την εξέταση των επιχειρησιακών προγραμμάτων γιατί είχε ήδη ευθυγραμμιστεί με τους στόχους για την πλειονότητα των στόχων έχουν γίνει κάποιες αλλαγές ως προς την χρηματοδοτική υποστήριξη βάσει κάποιων κριτηρίων που δεν έγιναν απολύτως σεβαστά. Στην επόμενη διαφάνεια, δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε πολύ καλά, Από την περίοδο ε, από το 7 ως το 13, των επιχειρηματικών προγραμμάτων από το 7 ως το 13, μπορείτε να δείτε ε, ότι σε γενικές γραμμές, εντάξει υπήρχαν κάποιες αδυναμίες, όμως ε, είναι από τις λίγες εκθέσεις μας, οι οποίες φαίνεται, φαίνονται πιο θετικά τα πορίσματα, είναι πιο θετικά από ότι τα αρνητικά ε, τα πορίσματα. Και βλέπουμε επίσης ότι ο ποσοστός ενσωμάτωσης των στόχων σε επιχειρησιακά προγράμματα είναι υψηλού επίπεδου, ε, για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 85%, 58% για την ε, τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως επίσης για τη λογική των εργαλείων παρακολούθησης που είναι βασικό στοιχείο. Ε, βλέπουμε ένα χαμηλό επίπεδο, ένα σχετικά χαμηλό επίπεδο επιχειρησιακών προγραμμάτων που, όπου δεν γίνεται αυτή η ανάλυση αναγκών. Για όσους ας πούμε εγκαταλείπουν το σχολείο νωρίς, μόνο το 4% απουσιάζει. Ε, Αποσκιάζει δηλαδή το, το, το πλαίσιο ε, ε, περιγραφής της κατάστασης Νομίζω όμως ότι είναι μάλλον θετικά και όχι αρνητικά τα απορέσματα. Επόμενη διαφάνεια. Μπορούμε να δούμε και να συγκρίνουμε την αξιολόγηση Τη κατάρτιση των επιχειρησιακών προγραμμάτων από το 2014 έως το 2020. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, καθοδήγησε τα κράτη-μέλη σε σχέση με την κατάρτιση αυτή. Τα προγράμματα ήταν συμβατά με τους στόχους της εκπαίδευσης της Ένωσης και επίσης ε, βρήκαμε και επαρκή περιγραφή της λογικής παρέμβασης και Επίσης, ε, υπάρχει ένα νέο βελτιωμένο νομοθετικό πλαίσιο. Παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμη δύο αδυναμίες. Το πλαίσιο δεν αναφέρει λεπτομερώς ε, τις ε, τους δείκτες που θα έπρεπε να ε, αξιολογούν την κάθε επένδυση και το αποτέλεσμα της. Ε, υπάρχει λοιπόν ε, μία έλλειψη συνέπειας μεταξύ των οπερισιακών προγραμμάτων. Επίσης δεν συνδέονται τα μέτρα εκπαίδευσης με τα μέτρα απασχόλησης. Δεν υπάρχει λοιπόν επαρκώς αυτός ο σύνδεσμος μεταξύ της εκπαίδευσης ε, και ε, της απασχόλησης. Η διαδικασία λοιπόν ε, εξέτασης των επιχειρησιακών προγραμμάτων δείχνει κάποια βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Το βασικό επόμενο βήμα που είναι η εφαρμογή επαφίεται στα κράτη-μέλη για να επιλέξουν και να εφαρμόσουν τα κατάλληλα προγράμματα για να επιτύχουν, να υποστηρίξουν την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Επόμενος πίνακας. Βλέπετε ότι ε, ότι είναι ακριβώς το ίδιο πλαίσιο με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, αλλά εδώ μπορείτε να συγκρίνετε, μπορείτε να συγκρίνετε τις σημαντικές βελτιώσεις ε, σε σχέση με την συμπερίληψη των στόχων των επιχειρησιακών προγραμμάτων για όσους εγκαταλείπουν το σχολείο νωρίς. 88% ε, κάλυψη και για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 63% και για την λογική παρέμβασης, ε, παρέμβασης και για τα εργαλεία παρακολούθησης βλέπουμε ότι περίπου ότι σχεδόν όλα καλύπτουν ε, τις ε, προϋποθέσεις και αυτό πραγματικά αποτελεί μία σημαντική βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Επίσης, η έκθεσή μας συμπεριλαμβάνει τέσσερις συστάσεις, ε, τις οποίες έχει αποδεχθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν εφαρμοστούν θεωρούμε ότι θα βελτιώσουν περαιτέρω την ε, ε, βελτίωση της εφαρμογής. Οι συστάσεις αυτές αφορούν τους δείκτες αποτελεσμάτων, τους ε, δείκτες παρακολούθησης ε, ε, αξιοποίησης των κονδυλίων επειδή είναι η νεολαία και η απασχόληση αναφέρθηκε πολλές φορές και το είπατε κι εσείς ότι ασχολείστε με αυτό το θέμα πολύ στην Επιτροπή σας κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι καλό είναι να πούμε επίσης ότι υπάρχουν τρεις εκθέσεις που αφορούν τους νέους και την απασχόληση. Η τρίτη δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί αυτή όμως είναι η πρώτη που δημοσιεύσαμε πριν ε, από ένα χρόνο περίπου σαν αφορά την εγγύηση για τους νέους και τα πρώτα ε, βήματα που έχουν γίνει για την εφαρμογή αλλά και τους ε, κινδύνους που μπορεί να προκύψουν. Αναλύσαμε τον σχεδιασμό των διαφόρων μέτρων των κρατών μελών σε σχέση με τους νέους και την απασχόληση και είδαμε ότι έχουν γίνει τα πρώτα βήματα. Πράγματι όμως εντοπίσαμε και τρεις βασικούς κινδύνους Όσον αφορά τώρα τα επαρκή κονδύλια, μερικά ακόμα αριθμητικά στοιχεία το ποσό χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμο, που ξέρουμε ότι είναι 12,7 δισεκατομμύρια για ολόκληρο, ολόκληρη την εγγύηση ε, για τους νέους, κάποιες ε, εκτιμήσεις από το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας ε, δείχνουν πολύ, πολύ υψηλότερα ποσά σε σχέση με τη χρηματοδότηση 21 δις ε, κατέτος είναι η, η εκτίμηση και είναι πολύ λιγότερο το ποσό, πολύ μικρότερο το ποσό που είναι διαθέσιμο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που διαπιστώσαμε, ο μεγαλύτερο κίνδυνο. Η χρηματοδότηση για την εγγύηση των νέων δεν είναι επαρκώ πρικοδοτημένη. Για κάθε νέο άνθρωπο που δεν συμμετέχει στην εκπαίδευση ή στην κατάρτιση. Επόμενο κίνδυνο είναι η έλλειψη κατάλληλου ορισμού τι θα πει ποιότητα. Γιατί η καλή ποιότητα σε ένα κράτο μέλο μπορεί να μην είναι καλή ποιότητα, ίδια, δεν είναι, μπορεί να μην, να μην είναι ορισμό ο ίδιο μεταξύ των ε, διαφορετικών κρατών μελών. Κάποιοι, α πούμε, θεωρούν η διάρκεια της ε, σύμβασης απασχόλησης ε, είναι το πιο χαρακτηριστικό κριτήριο. Άλλοι θεωρούν τον ελάχιστο μισθό. Φυσικά είναι πλήρης αρμοδιότητα των κρατών μελών και αποκλειστική ε, ορισμός αυτών των κριτηρίων, αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει να πιστεύουμε ότι αυτή η απουσία κοινού ορισμού όσον αφορά την ποιότητα της εργασίας είναι ένας κίνδυνος. Είναι ένας κίνδυνο. Τρίτος σημαντικός κίνδυνος που εντοπίσαμε και που δεν έχει να κάνει μόνο με την εγγύηση για τους νέους. Είναι γενικώ ένα πρόβλημα που ξέρουμε και από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και το προηγούμενο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι η παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων για τα εργαλεία. Και κάποιες πληροφορίες να σας γνωστοποιήσω ότι αυτή η τρίτη έκθεση για τους νέους και την εργασία που αξιολογεί τα αποτελέσματα σε επίπεδο κρατών μελών, τι, έχει επιτευχθεί δηλαδή από την εγγύηση των νέων, θα δημοσιευθεί στις 4 Απριλίου. Οπότε, μόλις δημοσιευθεί, βεβαίως εμείς θα σας την ε, διαβιβάσουμε, θα τη δημοσιεύσουμε και στον ιστότοπό μας και εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εμείς οργανώνουμε, σας προσκαλούμε, είστε όλοι ευπρόσδεκτοι, μία διάσκεψη για την απασχόληση των νέων εδώ, εδώ στο Κοινοβούλιο, στις 10 Μαΐου. Με πολύ χαρά θα περιμένουμε να σας δούμε εκεί όλους για να συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Ε, ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ε, εντυπωσιακή έκθεση. Και επίσης ευχαριστούμε πολύ που το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο προφανώς ε, ασχολείται εντατικά με τα θέματα αυτά και μπορεί να μας δώσει σημαντικές επισημάνσεις εν σχέση με το τι θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε να αλλάξουμε στην ε, δομή, στη διάφραση των προγραμμάτων. Ε, γιατί το γεγονός ότι περιορισμένη πόρ για όλα τα προγράμματα, αυτό το γνωρίζουμε όλοι, είναι κοινό τόπο, και εδώ γίνονται πολλές αντιπαραθέσεις με την Επιτροπή αλλά και τι χώρες μέλη και ίσω θα μπορούσαμε να σα ε, να δούμε ότι είναι σημαντικό το να επισημαίνει και το ελεγκτικό συνέδριο ότι ορισμένα προγράμματα υποχρηματοδοτούνται έχει άλλο κύρος το να το λέει το ελεγκτικό συνέδριο και είναι διαφορετικό όταν το λέει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχει πολιτικά ε, κίνητρα. Η Σαμπίνε, καταρχήν θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που είχαμε την παρουσίαση αυτή της έκθεσης εδώ εν συντομία Πιστεύω ότι θα είναι ασφαλώς ενδιαφέρον να δούμε τη δημοσίευση αυτή, νεότητα και απασχόληση, για να μπούμε στις λεπτομέρειες. Έγινε σαφές ότι υπάρχουν ε, ε, διαφορές μεταξύ της ε, προηγούμενης και της τωρινής περίοδου ισχύου των προγραμμάτων. Θα ήθελα να τονίσω το ότι είπε η Πέτρα προηγουμένως ότι με αυτά τα προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ε, δεν υπάρχουν αρκετοί πόροι. Τα προγράμματα αυτά υποχρηματοδοτούνται. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αν δεν υπάρξουν κονδύλια. Θα ήθελα και εγώ να το τονίσω. Και νομίζω ότι ένα σημαντικό μέλημα μελλοντικά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να υποστηριχθούν οι χώρες που υπάρχουν υψηλά ποσοστά ανεργία των νέων, ούτω ώστε να δημιουργηθούν κάποιε δομέ που να μπορέσουν να δώσουν, να εξασφαλίσουν λύσει στο πρόβλημα. Γιατί θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες προοπτικές ε, για αυτούς τους νέους. Ε, ίσως η ανταλλαγή των πρακτικών είναι ένας τρόπος και το πώς μπορούν να τέχουν εφαρμογή στο οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο μιας άλλης χώρας. Και αυτό είναι σημαντικό. Και εμένα θα με ενδιάφερε να έχουμε κάποια στιγμή κάποιες συγκριτικές ε, αξιολογήσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά την εγγύηση για τους νέους. Ε, το πρόγραμμα δεν πηγαίνει τόσο καλά σε χώρες που θα το είχαν κατεπηγόντως ανάγκη. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει επαρκέστερη ενημέρωση. Ε, πώς θα έχει το πρόγραμμα, γιατί και το ζητούμενο δεν είναι μόνο η αποτελεσματική ε, ε, χρήση των χρημάτων αλλά και το σε ποια κατεύθυνση πως ε, αποτιμάται αυτή η αποτελεσματικότητα θα πρέπει να συνδεθεί άμεσα με την απασχολησιμότητα. Ε, μπορούμε να δώσουμε πολλά χρήματα για το λάθος στόχο και λίγα χρήματα για κάτι που θα υπήρχε μεγαλύτερη ανάγκη. Ευχαριστούμε πολύ και εγώ από τη δική μου πλευρά θα ήθελα να υποβάλω ένα ερώτημα σε αντίστοιχη κατεύθυνση όπως και η συνάδελφος προηγουμένως ιδιαίτερα όσον αφορά τους νέους εμείς ως Κοινοβούλιο αρχικά υπήρξαμε κάπως ματαιωμένοι για το γεγονός ότι ήταν τόσο περιορισμένοι οι πόροι που είχαμε στη διάθεσή μας και είπαμε ότι χρειαζόμαστε τα τριπλάσια κονδύλια, αλλά τελικά υπογραφήκαμε στη τελική φάση να διαπιστώσουμε ότι τα χρήματα τελικά δεν ε, δόθηκαν ή δεν αξιοποιήθηκαν αποτελεσματικά γιατί οι χώρες ε, μέλη που τα χρειάζονται κατεπηγόντως δεν έχουν μια ιδέα του πώς να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα αυτά ούτως ώστε ε, να μπορέσουν ε, να υποφεληθούν από αυτά οι νέοι. Άρα η ορθή χρήση των ε, κονδυλίων αποτελεσματικά εις όφελος των νέων ανθρώπων. Και αν δούμε μία από τις πρώτες διαφάνειες που μας δείξατε, τα κονδύλια του ΑΕΣΕΦ ε, για τους νέους. Νομίζω ότι το ποστό αυτό έχει μειωθεί. Το τι επενδύουν οι χώρες μέλη. Αυτό αφορά το σύνολο της διάρκειας ισχύων των, προγρα... Ε, προγραμμάτων ή αφορά ε, το χρόνο που έχουν τρέξει μέχρι τώρα. Άρα λοιπόν μπορούμε να απομένουμε ότι τουλάχιστον στη συνέχεια θα φτάσουν στα ποσοστά στα οποία έλθαν τα προηγούμενα προγράμματα είναι μια πρόγνωση που αφορά τη συνολική διάρκεια ισχύω των πραγμα... προγραμμάτων. Πραγματικά είναι τρομερό, είναι τρομερή η διαπίστωση αυτής της μείωσης. Ο συνάδελφος κ. Βέντερ. Αν εφόσον μιλάμε γερμανικά, θα προσπαθήσω και εγώ να μιλήσω στα γερμανικά. Εδώ μιλάμε για την έκθεση αυτή που αφορά την παρούσα κατάσταση. Οι πληροφορίες είναι ότι υπάρχει μια μείωση, όπως είπες. Το θέμα είναι τι θα γίνει μελλοντικά. Χρειαζόμαστε και κάποια δεδομένα από τις χώρες μέλη. Κατά τα άλλα θεωρώ ότι ήταν ενδιαφέροντα τα όσα ακούσαμε. Ευχαριστώ. herzlichen Frau... Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ιβάνοβα, θέλετε εσείς να απαντήσετε και να δούμε κατά πόσα ανακύπτουν άλλα ερωτήματα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντικά τα ερωτήματα. Θα αρχίσουμε με το ερώτημα της κυρίας Φερχάη. Και εσείς μιλήσατε, κυρία Πρόεδρε, για τη χρηματοδότηση. Δηλαδή, στην ουσία μιλάμε για χρήματα. Υπάρχουν αρκετά χρήματα για να χρηματοδοτηθούν οι στόχοι που έχουμε ορίσει. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και στα πρώτα στάδια της χρήσης του, των, ε, του Ταμείου Εγγύσεων για τους ε, νέους. Δηλαδή, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε το, ε, το σχεδιασμό του προγράμματος για να δούμε τι γίνεται με τις έγκαιρες προειδοποιήσεις και τα απαγορευτικά για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε άμεσα για να βοηθήσουμε τους νέους για να βρούνε θέσεις εργασίας, να εκπαιδευτούν ή να καταρτιστούν. Και υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Στην έκθεση είπαμε ότι είναι ανεπαρκής η χρηματοδότηση. Ίσως μπορούμε να πούμε ότι ναι, δεν υπάρχουν χρήματα, για την ε, χρηματοδότηση αυτών των μέτρων ή με βάση τις ε, υποσχέσεις και τις υποχρεώσεις τα χρήματα δεν αρκούν. Γνωρίζουμε δηλαδή ότι η χρηματοδότηση είναι ελιπέστατη και είναι όλο ένα και πιο περιορισμένη. Άρα πρέπει να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα μέσα και στην έκθεση αναφέρουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη προτεραιότητα των μέτρων με βάση τα, τις ανάγκες και των κρατών μελών. Η, αυτό το, αυτή η εγγύηση για τους νέους, κάτι θα μας πει και η Κομισιόν, αλλά έχει δεμένα τα χέρια. Γιατί δεν μιλάμε για ένα νομοθετικό πλαίσιο κάλυψης, δεν υφίσταται κάτι τέτοιο, γι' αυτό τα κράτη-μέλη θα θέσουν προτεραιότητες ως προς τα μέτρα και θα χρησιμοποιήσουν τη, τους διαθέσιμους πόρους Ενδεχομένως, γιατί εάν δώσετε υποσχέσεις ότι θα βρείτε εργασία για κάθε νέο στην Ευρώπη, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το κόστος είναι υψηλό. Με την παρούσα χρηματοδότηση θεωρούμε ότι δεν μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες και οι επιπτώσεις τους. Η κυρία Φερχάιν μίλησε και για την ε, εκμάθηση, για τη μάθηση από τις βέλτιστες πρακτικές. Αυτό που προσπαθούμε είναι όχι μόνο να έχουμε μία δίκαιη αποτίμηση που ενέχει και θετικές επικρίσεις, αλλά να χρησιμοποιήσουμε και τις βέλτιστες πρακτικές. Γιατί θα πρέπει να μαθαίνουμε όχι μόνο από τα λάθη, από τα λάθη μας, αλλά και από τις βέλτιστες πρακτικές και παραδείγματα. Αυτό αναφέρεται και στην έκθεση βεβαίως. Σε αυτό το στάδιο δεν θα ήθελα να πω περισσότερα για την ε, τρίτη έκθεση που θα παρουσιαστεί στις 4 ε, Απριλίου σε σχέση με τα πραγματικά αποτελέσματα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η έκθεση, πολύ σημαντικά τα ευρήματα, αλλά δεν θα ήθελα να πω περισσότερα σε αυτό το στάδιο. Όμως υπάρχουν καλά παραδείγματα. Το δείγμα των κρατών είναι σκόπιμο, σκόπιμα επιλεγμένο για να δούμε πώς κράτη με υψηλό δίκτυ ανεργίας ε, μπορούν να παρέχουν βέλτιστες πρακτικές για άλλες χώρες. Και αυτό βέβαια βέβαια σχετίζεται με τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης, αλλά πιστεύω ότι αν μοιραστούμε αυτά τα στοιχεία βέλτιστων ε, πρακτικών, έχουμε να κερδίσουμε όλοι. Ο κύριος Βέντα μίλησε ε, για τα κράτη-μέλη. Γιατί αυτά τα συγκεκριμένα κράτη-μέλη, σας είπα στην αρχή ότι έχουμε μία σειρά κριτηρίων σε σχέση δηλαδή με τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων κρατών μελών και για τα κράτη που επιδιώκουν μία γεωγραφική δίκαιη κατανομή. Τα κράτη-μέλη μας δίνουν παραδείγματα όπου καταδεικνύουμε αυτό που θέλουμε, αλλά αυτό είναι και το πιο συχνό ερώτημα και στην ετήσια δημοσιονομική μας ε, δήλωση. Και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε ποια κράτη ε, έχουν δαπανίσει όχι μόνο για κατάρτιση και εκπαίδευση, αλλά για να δώσουν και σημαντικά παραδείγματα. Τώρα, σε σχέση με το ρυθμό δαπάνης, δαπανών, μιλάμε για 20,71 ε, δις και θα μας πει η Επιτροπή περισσότερα, αλλά αυτή ήταν η εικόνα που είχαμε σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. που και αυτά τα στοιχεία δείχνουν πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση, αλλά αυτό είναι προσωπική μου άποψη. Εάν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, έχω εγώ μία. Ασφαλώς, ε, εξετάσετε τι γίνεται με το ISF και τι επενδύεται από εδώ στο, για τους νέους. Εμείς είμαστε αρμόδιοι για το μεγάλο πρόγραμμα κινητικότητας ε, ε, Europe ε, Plus και για το πρόγραμμα Europe for Citizens. Όλοι ομοφωνούν λέγοντας ότι οι πόροι είναι περιορισμένοι. Σήμερα δεν θα ήθελα να μου απαντήσετε σε αυτό. Αυτό το οποίο κάναμε σήμερα για το ISF, ίσως ενδεχομένως θα μπορούσε να γίνει μελλοντικά για το Erasmus Plus και για τα δύο άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα, γιατί αυτό θα ήταν για μας χρήσιμο, θα μπορούσε να μας παράσχει χρήσιμες πληροφορίες, ιδιαίτερα όσον αφορά την μελλοντική περίοδο ισχύω των προγραμμάτων. και αν θέλουμε να δούμε τα πράγματα αντικειμενικά και αν είχαμε μία ένδειξη ότι πραγματικά έχουμε δίκιο ότι υποχρηματοδοτούνται τα προγράμματα και ότι θα χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι τους οποίους έχουμε διατυπώσει, θα ήταν χρήσιμο. Δεν χρειάζεται να απαντήσετε τώρα αυτή την ερώτηση. Μπορείτε να τη συζητήσετε με τους συναδέλφους σας κατά πόσο θα ήταν λογική αυτή η προσέγγιση. Αλλά για μας θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο εάν το ελεγκτικό συνέδριο ε, μπορέσει να το εξετάσει με μια κριτική ματιά. Και πραγματικά χαιρετήσουμε το γεγονός ότι ο ε, συνέδριο, ε, το ελεγκτικό συνέδριο δεν ε, προσλαμβάνει αυτόν σαν εκείνον ο οποίος ε, θέτει τον δάχτυλο επί των τύπων των ύλων, αλλά ε, θεωρεί αυτόν σαν ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κινηθούμε εξ αρχής προς τη σωστή κατεύθυνση και να μην είμαστε υποχρεωμένοι να αντιδρούμε εκ των υστέρων. όχι blaming και shaming, αλλά έγκαιρη προειδοποίηση και προβολή παραδειγμάτων ή μοντέλων που θα είχαν καλύτερα αποτελέσματα. Αν δεν θέλει να πάρει κανείς το λόγο, κύριε Βάνοβα, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε πράγματι είναι ένα κρίσιμο θέμα για το Εράσμος γιατί είναι πράγμα που είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους νέους ε, Youth Guarantee και εκπαίδευση είναι θέματα τα οποία μας απασχολούν πολύ και χαίρομαι που μπορώ να σας ενημερώσω ότι ήδη έχουν γίνει κάποια βήματα και κάνουμε έναν έλεγχο για το Erasmus Plus δεν μπορώ να πω ακριβώς πότε θα το ολοκληρώσουμε, αλλά θα διαβιβάσω ε, το μήνυμα συναδέλφους από την ενότητα 4, από, την, από το τμήμα 4, Chamber 4, και νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε μια αντικειμενική εικόνα όχι μόνο το κατά πόσο ένα, τα ποσά χρησιμοποιήθηκαν σωστά και χωρίς παρατυπίες, αλλά κατά πόσο ε, τα κονδύλια χρησιμεύουν ή εξυπηρετούν την επίτευξη των ε, δεδηλωμένων ε, στόχων. Ε, όπως είπατε πολύ σωστά, δεν θέλουμε να έχουμε μόνο το ρόλο του χωροφύλακα. Προσπαθούμε να είμαστε πιο αντικειμενικοί, επικοδομητικοί και να παράσχουμε έγκαιρες προειδοποίησεις. Γιατί πιστεύουμε ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από μία αντέδραση εκ των υστέρων. Για πράγματα που θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί εκ των προτέρων. Χαιρόμαστε λοιπόν γι' αυτό ε, και είμαστε στη διάθεσή σας για να σας υποβοηθήσουμε στην ε, βελτίωση των εκθέσεων. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και την παρουσία σας εδώ. Νομίζω ότι ήταν μια εξαιρετικά πολύτιμη συζήτηση. Μας δώσετε σημαντικές πληροφορίες και μας χαροποιεί ιδιαίτερα στο γεγονός ότι το ελεγκτικό συνέδριο ήδη εξετάζει το Erasmus Συν και αυτό θα μας βοηθήσει σίγουρα και γνωρίζω ότι στην, στο πεδίο της κοινή γνώμης αλλά και στο πολιτικό, στην πολιτική σκηνή τα ελεγκτικά συνέδρια θεωρούνται ως ε, χωροφύλακες γιατί ακριβώς θέτουν το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων. Αλλά μπορούν να λειτουργήσουν και πιο επικοδομητικά στο επίπεδο της πρόληψης και της έγκαιρης προειδοποίησης. Και αυτό μπορεί πραγματικά να μας βοηθήσει να κινηθούμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Σας ευχαριστούμε κυρία Ιβάνοβα. Είστε πρόσδεκτοι ανα πάσα στιγμή και καλή επιτυχία στις εργασίες σας. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, Αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα θα έρθουμε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασής μας και εδώ έχουμε πολλά χαρτιά και εδώ πρόκειται για τις μειονοτικές γλώσσες και την εκπαίδευση. Βέλτιστες πρακτικές και έχουμε μία παρουσίαση του Policy Department που πάντοτε μας είναι εξαιρετικά χρήσιμο παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες για την εργασία μας. Τον Ιανουάριο του 2016 η Επιτροπή μας είχε αποφασίσει να παρακαλέσει την ε, ε, μονάδα έρευνας να εκπονήσει μια μελέτη για τις μειονοτικές γλώσσες και την εκπαίδευση. Η έρευνα αυτή έχει ολοκληρωθεί ε, και χαίρομαι εκ των προτέρων για την ε, παρουσίαση. Ε, καλωσορίζω την κυρία Μέρκ από το Κέντρο Πολυγλωσσίας, η οποία θα μας παρουσιάσει τα σημαντικότερα ευρήματα. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε και έχετε το λόγο για 15 λεπτά επίσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισήγησή σας. Ε, ονομάζομαι Στέρκ και ασχολούμαι ε, στο κέντρο, απασχολούμαι στο κέντρο για τις ε, μειονοτικές γλώσσες και την εκπαίδευση και ε, συνεργάζομαι με τους Ντόμορα και Βαντεμίρ θα ήθελα λοιπόν να σας μιλήσω για την έκθεση αυτή. Θα σας πω, θα σας δώσω ορισμένα στοιχεία σε σχέση με το περιεχόμενο της έκθεσης. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να λάβουμε υπόψη ότι το 87 άρχισε αυτή η πολιτική και αυτό που μας ε, ενδιέφερε ήταν ε, η πολυγλωσία καθώς και οι μειονοτικές γλώσσες. Και τότε ψηφίστηκε μία πρόταση ψηφίσματος με ένα ξεχωριστό προϋπολογισμό για τις ε, μειονοτικές γλώσσες όμως το 2007 σταμάτησε αυτή η χρηματοδότηση και το Μέρκατον έγινε ένα κέντρο πληροφοριών και έρευνας που χρηματοδότησε η περιοχή του Φρίσλαν. Πρόκειται για έναν ανεξάρτητο οργανισμό έρευνας και θέλουμε η Φρίσλαν να ενταχθεί στην Ευρώπη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Προσπαθούμε να διαδώσουμε πολλές ε, πληροφορίες διασυνοριακά και γι' αυτό οι βασικές ε, δραστηριότητες του Μερκατόρ είναι να λάβει υπόψη την πολυγλωσία και την εκπαίδευση παντού στον ε, πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα και αυτό που έχει σημασία είναι και ο ρόλος των ΜΜΕ και πώς ε, χρησιμοποιούνται οι μειονοτικές γλώσσες και στα μέσα ενημέρωσης. Έχουμε συμμετάσχει σε πολλά σχέδια όπως το δίκτυο Mercator καθώς και σχέδια που σχετίζονται με τις γλώσσες των μεταναστών. Ε, έχουμε μία ε, ιστοσελίδα εμπεριστατωμένη για να δείτε τη δραστηριότητα του Μερκατόρ και έχουμε 600 εμπειρογνώμονες επιτόπου που ασχολούνται με την πολυγλωσία και την γλωσσική εκπαίδευση. Οργανώνουμε σεμινάρια για τις μειονοτικές γλώσσες που είναι γνωστά στην Ευρώπη και αλλού και η βασική μας εργασία αφορά την οριοθέτηση της εκπαίδευσης ως προς τις μειονοτικές γλώσσες από το Δημοτικό μέχρι το Πανεπιστήμιο. Έχουμε, τώρα διανύουμε τον πέμπτο χρόνο Μπορείτε να βρείτε όλα αυτά τα στοιχεία στην ιστοσελίδα που ενημερώνεται κάθε 10 χρόνια και είναι διαθέσιμα σε όλους. Και εκεί έχετε πολλές πληροφορίες για τις ε, μειονοτικές γλώσσες και την εκπαίδευση. Ε, έχουμε και το ε, μηνιαίο δελτίο τύπου Πέρσι το Σεπτέμβριο λάβαμε ε, ένα ερώτημα από την Επιτροπή σας να προβούμε σε μία εις βάθος ανάλυση για τις μειονοτικές ε, γλώσσες, την εκπαίδευση, δηλαδή τη δυνατότητα των μειονοτήτων να εκφραστούν στη μητρική τους ε, γλώσσα. Να έχουμε δηλαδή τους δείκτες για τις μειονοτικές γλώσσες έτσι ώστε να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε το μη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης υπήρχαν ε, και στοιχεία για τους πτυχιούχους που χρησιμοποιούσαν μειονοτικές γλώσσες και πώς μπορούν να επανενταχθούν στις κοινότητές τους. Ήταν λοιπόν ε, ένα εμπεριστατωμένο ε, θέμα και ερώτημα ασχοληθήκαμε με 13, ε, ε, με 13 υποθέσεις και περιπτώσεις μέσα στα πλαίσια τη Μερκατόρ και αυτά τα στοιχεία μπορούσατε να τα βρείτε στα, στους φακέλους μας. Λάβαμε συνεντεύξεις και επίσης Είδαμε ποια είναι η τεκμηρίωση στον τομέα και ποιες συστάσεις ήδη υπήρχαν στο παρελθόν που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Αυτές οι κατά περίπτωση μελέτες ήταν και η πεντουσία των ερευνών. Κάναμε μια συγκριτική μελέτη Είδαμε όλες τις ε, κατά μελέτες και τις εντάξαμε στην, ε, στην ανάλυση, στη συγκριτική αυτή ανάλυση. Και όπως ε, σας είπα, ασχοληθήκαμε με 13 περιπτώσεις που τις βλέπετε στη διαφάνεια πίσω μου. Δεν θα ήθελα να τις κατονομάσω όλες τις περιπτώσεις μπορείτε να ε, κοιτάξετε τους φακέλους, να τους συμβολευτείτε όποτε επιθυμείτε. Ένα από τα πρώτα ζητήματα στην ερευνητική πορεία είναι η ορολογία που χρησιμοποιείται. Ε, δηλαδή εγώ όταν ε, λέω τυρί σκέφτομαι το τυρί γκούντα, ενώ για έναν Γάλλο το τυρί είναι το καμαμπέρ. Δηλαδή ο καθένας έχει διαφορετικές εικόνες ε, κατά νου σε σχέση με ένα συγκεκριμένο προϊόν και αυτό αφορά και τις μειονότητες. Ένας άλλος παράγων είναι ότι δεν υπάρχει ένας συμφωνημένος όρος για το τι σημαίνει μειονότητα. Γι' αυτό χρησιμοποιήσαμε τον όρο που υπάρχει στον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις μειονοτικές γλώσσες, δηλαδή τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά σε ένα συγκεκριμένο έδαφος ή εδαφικό διαμέρισμα ενός κράτους, όπου ζουν μειονότητες ή αυτόχθονες πληθυσμοί. Δεν μιλήσαμε δηλαδή, δεν ασχοληθήκαμε με τις νέες μειονότητες, δηλαδή τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που διαβίουν σε μια συγκεκριμένη χώρα. Ε, έχω ένα μικρό βίντεο ε, από το κέντρο Μαρίσκο το οποίο δείχνει ποια είναι τα δικαιώματα των μειονοτήτων και γιατί θέλουμε να τις ε, προστατεύσουμε. Θα ήθελα να σας δείξω αυτό το βίντεο εάν ε, λειτουργεί το σύστημα. Στο δικό μου υπολογιστή λειτουργεί μια χαρά αλλά εδώ βλέπω ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Όταν δείτε τι γίνεται το, με το Ευρωπαϊκό Κέντρο ε, Θεμάτων Μειονοτήτων, μπορείτε να δείτε να κάνετε αυτή την προβολή μόνοι σας. Ως προς το θεωρητικό μας πλαίσιο, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, και νωρίτερα, οι διεθνείς οργανώσεις προέβαλαν πρότυπα και μηχανισμούς για την προστασία των μειονοτήτων και οι μειονοτικές γλώσσες εντάσσονται στην πολιτισμική ε, ποικιλότητα, όπως ισχύει και με τη βιοπικιλότητα. Ένα άλλο θέμα αφορά τις εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες για να φτάσουμε σε μια πιο ειρηνική και σταθερή Ευρώπη. Άρα ο στόχος είναι η ειρήνη στην Ήπειρο. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει συντάξει δύο διεθνείς συνθήκες για την προστασία των μειονοτικών γλωσσών, ο Ευρωπαϊκός Χάρτης για τις μειονοτικές γλώσσες και το πλαίσιο, η σύμβαση πλαίσιο για την προστασία των μειονοτήτων. Αν δεν γνωρίζετε ε, τον χάρτη μπορώ να σας τον εξηγήσω κατά τη διάρκεια των ερωταποκρίσεων. Και η διαφορά μεταξύ των δύο είναι ότι ο Ευρωπαϊκός Χάρτης προστατεύει μειονοτικές γλώσσες, ενώ η Διεθνή Σύμβαση προστατεύει πρόσωπα που ανήκουν σε μειονότητες. Ε, με βάση την αρχή της επικουρικότητας, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν λίγο επιφυλακτική ως προς τον παρεμβατισμό, την παρέμβαση για θέματα μειονοτήτων, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια έχουν αναλυφθεί αρκετές πρωτοβουλίες σε σχέση με περιφερειακές μειονότητες και τα γλωσσικά τους δικαιώματα. Ένα από τα θέματα που θα ήθελα να τονίσω είναι το ψήφισμα για τις μειωτικές γλώσσες που κινδυνεύουν. Ο Φρανσουά Αλφόνση ε, συνέταξε αυτή την έκθεση και εγκρίθηκε με κατά 92% αυτό το 2013. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο έκτοτε έχουν ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα για να τεθεί στην πράξη το ψήφισμα αυτό. Σας μίλησα για την ιστοσελίδα μας, ε, για την, ε, τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Μειωτικών Γλωσσών και την ε, Σύμβαση Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις μειονότητες. Υπάρχουν πολλές εκθέσεις και τεκμηρίωση. Υπάρχουν, ξέρετε ποιες είναι οι χώρες που έχουν κυρώσει και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη και την, ε, το πλαίσιο, τη συμφωνία πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας. Ως προς την έκβαση τώρα και την ολοκλήρωση των εκθέσεων, σας είπα ότι έγινε μία συγκριτική μελέτη με βάση 13 περιπτώσεις και ε, λάβαμε υπόψη μια συγκεκριμένη πλαισίωση μελετών για κατά περίπτωση μελέτες, αλλά στο τομέα της εκπαίδευσης δεν ήταν δυνατόν να συγκρίνουμε τις ε, επιμέρους περιπτώσεις. Γι' αυτό προσπαθήσαμε να βρούμε συσχετισμούς, δηλαδή ε, προκλήσεις ή ε, βέλτιστες πρακτικές που αντιμετωπίζουν οι μειονότητες. Και εντάχει θα σας μιλήσω για αυτά τα σημεία που βλέπετε επί της οθόνης. Ένα από τα βασικά στοιχεία είναι το καθεστώς επίσημης γλώσσας. Όπως σας είπα, δεν υπάρχει συμφωνημένος ορισμός για τις μειονότητες, αλλά σε κάθε χώρα αντιμετωπίζεται ίσως κάπως διαφορετικά η μειονοτική γλώσσα. Ας πούμε στην Ιρλανδία εμείς λέμε ότι είναι μειονοτική γλώσσα, αλλά στην Ιρλανδία είναι η πρώτη επίσημη γλώσσα του κράτους. Άρα η κατάσταση είναι διαφορετική στη βασική χώρα δηλαδή ή στην Ουαλία, γιατί η, η γλώσσα αυτή είναι η πρώτη της ε, αυτόνομης κοινότητας. Και αυτό αφορά και τα σερβικά, που έχει ένα συγκεκριμένο καθεστώς στη, στην, στον Ευρωπαϊκό Χάρτη. Και σας τα λέω αυτά γιατί υπάρχει διαφορά ως προς το καθεστώς αντιμετώπισης της γλώσσας, κατά πόσο είναι μειονοτική γλώσσα ή επίσημη γλώσσα, επίσημη γλώσσα του κράτους ή της περιοχής. Σας μίλησα για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη και την Σύμβαση Πλαίσιο και ε, οι δύο αυτές ε, συνθήκες ή συμβάσεις είναι οι πιο γνωστές γιατί προβλέπουν και ένα σύστημα ελέγχου για να υπενθυμίσουμε σε όλους τι είναι οι μειονότητες, Γι' αυτό θα πρέπει τα κράτη να έχουν κυρώσει αυτές τις δύο συμβάσεις. Αλλά δεν είναι και προαπαιτούμενο αυτό, γιατί στη Νότια Ευρώπη, ας πούμε, η, η Ιταλία υπέγραψε τη σύμβαση, αλλά δεν την κύρωσε. Άρα ε, θα πρέπει να δούμε σε αυτή την περίπτωση τι θεωρείται ευέλτιστη πρακτική. Άρα η υπογραφή ε, των δύο αυτών πράξεων δεν είναι ε, πρόκριμα για τις ε, καλές πρακτικές. Επίσης, αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε κατά πόσο μία μειονότητα παραμένει σε μία συγκεκριμένη εδαφική ε, ενότητα η περιοχή, όπως ε, ισχύει στις περιπτώσεις των γερμανικών ομόσποδων ε, κρατηδίων στη Φρισλάνδη. Ε, ισχύει κάτι τέτοιο. Στην περίπτωση της Ρουμανίας είναι εντελώς διαφορετικό γιατί η μειονότητα, η ουγγρική μειονότητα δεν μπορεί πάντα να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα της ως προς ε, το να εκφραστεί προς τις δημόσιες αρχές. Και αυτό που έχει σημασία είναι ο ρόλος του κράτους. Πώς αντιμετωπίζει τις γλώσσες γιατί ένα κράτος μπορεί να ενισχύσει ή να καταρακώσει μία μειονότητα. Βλέπουμε λοιπόν τι γίνεται συγκεκριμένο προς τις νομοθετικές πράξεις από τα διάφορα κράτη-μέλη. Γιατί οι Ούγγροι στη Σλοβακία ε, στη Ρουμανία ε, μπορούν να έχουν υποστήριξη από την Ουγγαρία, γιατί πρόκειται για όμορες χώρες. Όταν ε, μιλάτε για την Ουαλία, στην περίπτωση της Ουαλίας, αυτό που έχει σημασία είναι ποια είναι η κρατική πολιτική έναντι των μειονοτήτων. Γλωσσικός προγραμματισμός. Ε, έχει μεγάλη σημασία γιατί χορηγούμε δικαιώματα στις μειονότητες, το δικαίωμα στην εκπαίδευση, αλλά αν δεν εφαρμοστεί είναι κενό γράμμα. Άμα πείτε ότι είμαι από τη Φρίσλανδ, γνωρίζω αυτή την περίπτωση, και δικαιούμε εκπαίδευση στο σχολείο, αυτό ισχύει θεωρητικά. Ε, η κόρη μου είναι 4 χρονών που πηγαίνει σχολείο στο πολύ, ε, πολύ κοντά στο σπίτι μας, στην κοινότητά μας, στη μικρή μας κοινότητα, αλλά ε, δυστυχώς ε, διδάσκεται μόνο Ολλανδικά. Άρα έχει μεγάλη σημασία ο γλωσσικός προγραμματισμός. Δεν μιλάμε μόνο για την εκπαίδευση, αλλά και διάφορους τομείς, επιμέρους τομείς. Πώς μπορούν να κατανοήσουν οι άνθρωποι τα πλεονεκτήματα της πολυγλωσσίας, ότι έχει μεγάλη σημασία να μιλούν μια μειονοτική γλώσσα. Πώς ε, οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια μειονοτική γλώσσα επικοινωνιακά ή στον τομέα υγείας, πώς να αναγνωρίσουν υπεύθυνοι τη σημασία της γλώσσας, της χρήσης μιας μειονοτικής γλώσσας από τους νοσηλευτές, ας πούμε. Γι' αυτό ο γλωσσικός προγραμματισμός έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή έχει σημασία να δούμε πώς μπορούν να εφαρμοστούν αυτά τα δικαιώματα που υπάρχουν στο γράμμα του νόμου. Ως προς τα εκπαιδευτικά πρότυπα, είδαμε για τις βέλτιστες πρακτικές και Μιλάμε για την ε, ε, εκπαίδευση σε δύο γλώσσες. Ας πούμε στη βασκική χώρα χρησιμοποιούνται και τα ισπανικά και τα αγγλικά παράλληλα με τα βασκικά. Και υπάρχουν και ε, σχολεία που χρησιμοποιούν δύο γλώσσες. Αλλά δεν υπάρχει ένα μέτρο για όλους. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα πρότυπο τριών γλωσσών έφνη σε όλα τα σχολεία. Θα πρέπει να βρούμε τις, ε, να αποτιμήσουμε τις επιμέρους καταστάσεις, τι ισχύει στις περιφέρειες και ούτω καθεξής. Δηλαδή γενικά θα πρέπει να δούμε ποιο εκπαιδευτικό πρότυπο θέλουμε να εφαρμόσουμε. Έχουμε την εθνική μας γλώσσα, αλλά θα θέλαμε να λάβουμε υπόψη και μία μειονοτική γλώσσα. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα σχήμα εθνικής επινόησης εκπαιδευτικού συστήματος. Ναι, θα επιταχύνω, νομίζω ότι επιβάλλεται. Μίλησα για την ευαισθησία όπως ε, όσο αφορά θέματα πολυγλωσσίας. Η πολυγλωσία πολλές φορές μπορεί να γίνει φόρτος αντί για πλεονέκτημα. Και σε όλες τις κατά περίπτωση μελέτες είδαμε ότι θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ένα ποιοτικό υλικό για την εκπαίδευση και φυσικά και εξειδικευμένο ε, διδακτικό προσωπικό για τις μειονοτικές γλώσσες που έχουν τη μειονοτική γλώσσα ως μητρική. Δυστυχώς, σε ορισμένα επαγγέλματα δεν χρησιμοποιούνται μειονοτικές γλώσσες όπως τη δημόσια διοίκηση ή στα νοσοκομεία από το νοσηλευτικό προσωπικό. Όταν προετοίμαζα αυτή την ε, παρουσίαση, σκεφτόμουν πώς θα ήταν μια ιδεώδης κατάσταση, χωρίς να αναφερθώ σε χώρες συγκεκριμένα. Είδαμε λοιπόν ότι εξελίχθηκαν πολλές ε, ε, χώρες στη χρήση μειονοτικών γλωσσών και εκεί που υπάρχει διοικητική αυτονομία υπάρχει μεγαλύτερη χρήση όπως Ουαλία ή η Βασκική χώρα. Αυτή είναι η καλύτερη πρακτική. Επίσης το κράτος πρέπει να έχει θετική στάση και να υπάρχει και χρηματοδότηση της ε, πολύγλωσσης εκπαίδευσης με διδακτικό προσωπικό και φυσικά ο μακροχρόνιος ε, προγραμματισμός έχει σημασία. Οι μειονοτικές γλώσσες πρέπει να χρησιμοποιούνται από, ήδη από την ηλικία του νηπιαγωγείου. Να βρούμε ένα επενδυτικό πρότυπο το οποίο να λειτουργεί σε επιμέρους περιφέρειες και να υπάρχει και ένα ε, σύστημα απτών, του κέρδους αυτών που χρησιμοποιούν τις ε, μειονετικές αυτών που χρησιμοποιούν τις μειονετικές γλώσσες. Η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι ποια είναι λιγότερο ιδεατή κατάσταση για τις μειονότητες. δηλαδή σε σχέση με μία χώρα όπου μιλείτε μία γλώσσα. Και αυτό που έχει σημασία είναι να λάβουμε υπόψη την γλωσσική ποικιλομορφία και αυτό σε χώρες όπου υπάρχει σταθερότητα, δηλαδή οι μειονότητες θα πρέπει να αναγνωρίζονται νομικά, εκπαιδευτικά και ούτω καθεξής. Δηλαδή δεν πρέπει μια χώρα να θεωρεί μια μειονοτική γλώσσα ως απειλή για τη χώρα ή να γίνονται διακρίσεις κατά των μειονοτήτων. Ή εκεί που δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση, δυστυχώς οι μειονοτικές γλώσσες δεν χρησιμοποιούνται. So then eh, θα επισπεύσω κάπως. Ας αφήσω την προγενέστερη διαφάνεια και ας σε αυτήν που βλέπετε. Τι θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπετε πολλές συστάσεις και συμπεράσματα στην έκθεσή μας. Αλλά εσείς είσαστε οι εμπειρογνώμονες ή και εσείς, γι' αυτό μπορείτε να λάβετε υπόψη συγκεκριμένε δράσεις. Θα πρέπει να ε, διατηρήσουμε και να προωθήσουμε προγράμματα που να σχετίζονται με την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών. Οι περιφέρειες θα πρέπει να μάθουν η μία από την άλλη, γι' αυτό χρειάζονται, χρειάζεται ανταλλαγή απόψεων και βέλτιστων πρακτικών, όπως προείπα. Και θα πρέπει να βοηθήσουμε οι μεν τους δε. Θα πρέπει να προωθήσουμε βοηθούσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση συστήματα εκμάθησης γλωσσών μέσα στα πλαίσια της πολυγλωσσίας. Και επειδή έχουμε όλο ένα και περισσότερους μετανάστες και πρόσφυγες, αυτό ε, αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία. Επίσης, το διδακτικό προσωπικό, η τεκμηρίωση έχει μεγάλη σημασία. Πολλές φορές οι μειονότητες είναι μικρές και είναι δύσκολο να εκδοθούν βιβλία στη γλώσσα τους. Επίσης, να προωθήσουμε σταθερές σχέσεις μεταξύ χωρών. Έτσι αναγνωρίζονται οι μειονότητες κάθε χώρας και να προωθήσουμε ένα διεθνές σύστημα ε, ευεργεσίας ή ευεργέτησης των μεν από τους δε και να προωθήσουμε μια ευρωπαϊκή ευαισθητοποίηση για την ε, πολυγλωσία. Γιατί σε πολλές χώρες υφίσταται η πολυγλωσία, αλλά θα πρέπει να προωθηθεί περαιτέρω. Σε άλλες χώρες η χρήση μειωτικών γλωσσών θεωρείται απειλή όμως να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να τους δώσουμε κίνητρα έτσι ώστε να ακυρώσουν και τις δύο συμβάσεις, άρα να συνεργαστούμε περισσότερο με το Συμβούλιο της Ευρώπης επί των θεμάτων αυτών. Επίσης να υπάρχει μακροχρόνιος γλωσσικός προγραμματισμός. Είναι κάτι που δεν ε, τελειώνει σε τρία-τέσσερα χρόνια γιατί τα πράγματα αλλάζουν με αργούς ρυθμούς και να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν τις μειονοτικές γλώσσες ήδη από το νηπιαγωγείο μέχρι και το πανεπιστήμιο. Ναι, μάλλον πρέπει να τελειώνω, έτσι δεν είναι. Ναι, λέει η Πρόεδρος, πράγματι. Κάτι το επιπρόσθετο. Ε, μίλησα για πληθώρα συστάσεων, μερικές έχουν τεθεί σε εφαρμογή, άλλες εντάσσονται στο, στο ψήφισμα του συναδέλφου σας. Δεν είναι κάτι το καινούριο. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι η εφαρμογή των μέτρων. Δεν μιλάμε μόνο για θεωρητική χορήγηση ορισμένων δικαιωμάτων. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να πιεστούν να θέσουν σε εφαρμογή αυτά τα νομοθετήματα. Αυτά είναι τα βασικά μου μηνύματα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ιόβια υπομονή σας. Αν ε, έχετε ερωτήσεις, με πολύ χαρά να σας απαντήσω. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν λίγο μακροτενέστερο από ό,τι είχαμε προβλέψει. Ευχαριστούμε πολύ για την ε, παρουσίαση της ε, μελέτης σας. Ο κύριος Σούγκορ. Ε, θα μιλήσω στα αγγλικά. Οι γλωσσικές μειονότητες είναι το 10% του πληθυσμού. Ωστόσο, τα... υπάρχουν ακόμα προβλήματα αναγνώριση εκ μέρου των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων το οποίο δείχνει ότι σε πολλές ε, χώρες ε, υπάρχουν προβλήματα. Για παράδειγμα η Ουγγρική μειονότητα στη Ρουμανία η οποία έχει 1,2 εκατομμύρια ανθρώπους. Ε, χάρηκα πάρα πολύ που ξεκίνησε μία μελέτη για την εκπαίδευση των μειονοτικών γλωσσών στην Ευρώπη. Ε, πάντως ε, η κατάσταση στην ε, Ρουμανία... Πάντω υπάρχουν κάποια σφάλματα όσον αφορά την κατάσταση στην Γερμανία. Και θα ήθελα να αναφέρω μια φράση για παράδειγμα. Στη σελίδα 26 το 7 το πιο σημαντικό πλεονέκτημα του να υπάρχει εκπαίδευση στην ουγγρική γλώσσα είναι ότι κανείς μπορεί να υποβάλει μια έτσι για εργασία στα ουγγρικά. Ε, και θεωρώ ότι αυτό δεν είναι ορθό γιατί το δικαίωμα εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα είναι θεμελιώδης ανθρώπινο δικαίωμα και διαφυλάτει το δικαίωμα των μειονοτήτων ε, στη γλώσσα τους και στην, ε, ως θεματοφύλακα της περαιτέρω ύπαρξής τους. Όλοι οι πολίτες, είτε είναι Ούγγροι είτε Ρωμά, έχουν το δικαίωμα να εκπαιδευεύονται στην ε, γλώσσα τους. Όσον αφορά τα επαγγέλματα στη Ρουμανία, για ανθρώπους που έχουν ε, σπουδάσει εκεί, συμφωνώ ότι είναι προς όφελος των μειονοτήτων, βεβαίως, να μάθουν τις μειονοτικές γλώσσες. Παρ' όλα αυτά, το κράτος θα έπρεπε να διευκολύνει ανθρώπους από άλλες ε, γλωσσικές προελεύσεις να διδάσκονται στη δική τους γλώσσα και όχι σύμφωνα με το σχολικό πρόγραμμα της πλειοψηφικής γλώσσας. Ε, ε, είναι μια γελία πλούστευση να πούμε ότι κάποιος ο οποίος διδάσκεται στα Ουγγρικά μπορεί να εργαστεί στην Ουγγαρία. Όσον αφορά τη Σλοβακία θα ήθελα να, ε, να διαβάσω δύο δηλώσεις στη σελίδα 1, Παρόλο που οι περισσότεροι ε, από την ε, μειονότητα οι περισσότεροι αναθρέφουν τα παιδιά τους στα Ουγγρικά και παρόλο που τα ε, και, και αυτό ακούγεται σαν οι γονείς οι οποίοι θέλουν να μεγαλώνουν στα παιδιά τους ε, σε ένα περιβάλλον ε, μειονοτικής γλώσσας, τη γλώσσα των γονέων, αυτό είναι αναχρονισμός. Και θεωρώ ότι θα έπρεπε να αποφύγουμε να γίνονται τέτοιου είδου ε, συμπεράσματα, γιατί όλοι έχουν το δικαίωμα να εκπαιδεύονται στη μητρική τους γλώσσα. Υπάρχουν πολλά μικρά, μικροσφάλματα, για να είμαι ευγενής θα το διατυπώσω έτσι. Έχω συντάξει ένα μακρύ κατάλογο. Ίσως θα μπορούσατε να τα διορθώσετε γιατί είναι απογοητευτικά. Köszönöm szépen. Mint a kezdeményezője a tanulmánynak, nagyon örülök. Ευχαριστώ. Εγώ πήρα την πρωτοβουλία της μελέτης αυτή. És και χαίρομαι πάρα πολύ. Εγώ την περίμενα αυτή τη μελέτη και επειδή αυτό το θέμα δεν λαμβάνει ιδιαίτερη προσοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά το γεγονός ότι εκτός από τις 24 επίσημες γλώσσες σύμφωνα με τις στατιστικές υπάρχουν έξι γλώσσες 79 ε, σύμφωνα με τη χάρτα δεν πρέπει λοιπόν να υποτιμούμε τη σημασία των γλωσσών αυτών, των μειονοτικών. Πρέπει οπωσδήποτε να ασχοληθούμε με αυτές. Όσον αφορά τώρα την ε, μελέτη που μόλις μας παρουσιάσατε, ε, με απογοήτευσε λιγάκι η μελέτη, γιατί όταν εγώ πήρα την πρωτοβουλία ο στόχος μου ήταν να ε, αναφέρεται κυρίως ότι η εκμάθηση μιας μειονοτικής γλώσσας είναι μια προϋπόθεση για την επιβίωση αυτής της γλώσσας, όμως νομίζω ότι ε, η έμφαση δίνεται σε κάτι διαφορετικό στη συγκεκριμένη μελέτη. Ο, το θεματικό τμήμα δεν ήρθε ποτέ σε επαφή μαζί μας. Με μας τους ευρωβουλευτές που πήραμε την πρωτοβουλία για τη μελέτη αυτή. Οπότε για μένα η μελέτη ε, δεν ε, παρουσιάζει τίποτε το καινούριο και επιπλέον έχει και πολλά σφάλματα, είδα πάρα πολλές αντιφάσεις στη συγκεκριμένη μελέτη. Διαβάζω ας πούμε ότι δεν υπάρχει πανεπιστήμιο ουγγρικής γλώσσας στη Σλοβακία, αλλά μετά ε, μία παράγραφο παρακάτω λέει ότι υπάρχει ένα πανεπιστήμιο. Κοιτάξτε, έχω πάρα πολλές, ε, πάρα, πολλά, ε, πάρα φορές διορθώσει διάφορα γραπτά κείμενα ε, και πρέπει να σας πω ότι απογοητεύομαι κάπως γιατί νομίζω ότι οι εμπειρογνώμονες με τους οποίους ήρθατε σε επαφή δεν ήταν οι κατάλληλοι. Δεν καταλαβαίνω γιατί ε, πήγατε για παράδειγμα ε, στο Άμστερνταμ να ρωτήσετε για τους Ούγκρους που ζουν στη Σλοβακία. Είναι προφανές ότι υπάρχουν και άλλοι εμπειρογνώμονες στους οποίους θα μπορούσατε να είχατε μιλήσει. Ε, ίσως θα, μπορείτε, θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε λίγο περισσότερο για ποιο λόγο ακολουθήσατε αυτήν την οδό. Πρέπει να πω ότι πολλά εξαρτώνται από τα κράτη-μέλη. Αν αυτές οι μειονοτικές γλώσσες ε, αποτελούν ε, μια αξία, ε, έχουν μια αξία για το συγκεκριμένο κράτος, τότε το κράτος θα υποστηρίξει την εκμάθηση των γλωσσών αυτών. Αν όχι, αν είναι διαφορετική η θέση του κράτους μέλους, η κατάσταση είναι εντελώ διαφορετική. Ε, νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα εάν τα σχόλια τα οποία μόλις έγιναν θα μπορούσαν να διαβιβαστούν στη γραμματεία και αντιστοίχως να διαβιβαστούν. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να υπησέλθουμε σε κάθε λεπτομέρεια. Βεβαίως υπάρχουν διαφορετικές ε, αξιολογήσεις για το ένα ή το άλλο σημείο, αποτιμήσεις. Δεν νομίζω θα πρέπει να δικολουθούμε και την κάθε φράση που συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση. Ίσως θα ήταν πιο φρόνιμο να υποβληθούν τα σχόλια και να δούμε πώς θα τα ε, συμπεριλάβουμε στην έκθεση. Παρακαλώ να είστε σύντομοι. Um, yeah, make it, um, very... Θα είμαι πολύ σύντομη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας. Έχουμε επίγνωση ότι ίσως ε, όλοι οι, όσοι πληροφορίες δεν είναι ορθές, ιδιαίτερα όταν κανείς ε, διαβάζει για τη χώρα του. Τα ντοσία αυτά ενημερώνονται κάθε 10 χρόνια. Έτσι λοιπόν οι πληροφορίες ε, αλλάζουν και πάντοτε προσπαθούμε να συμπεριλάβουμε αυτές τις πληροφορίες και να τις ελέγξουμε από ανθρώπους που γνωρίζουν καλώς την κατάσταση. Ε, έχουμε, θα εξετάσουμε 13 ε, περιπτώσεις ε, όπως σας είπαμε ε, και είναι, βέβαια, είναι πολύ δύσκολο σε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα να έχουμε τις εκτιμήσεις όλων των εμπειρογνωμόνων και να επικαιροποιήσουμε όλες τις πληροφορίες. Ε, είναι πολύ... Θα χρειαζόντουσαν τέσσερα χρόνια για να επισκεφθούμε όλες τις χώρες και να επαληθεύσουμε τα στοιχεία. Στο περιορισμένο χρονικό διάστημα που έχουμε στη διάθεσή μας κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά δύσκολο. Παρ' όλα αυτά είμαι ευτυχής για τα σχόλιά σας. Και αν ε, έχετε κάποιους εμπειρογνώμονες, είμαστε ευτυχείς να τους δεχτούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και για την επισήμανση που νομίζω ήταν σημαντική ότι αυτή δεν ήταν μια μελέτη η οποία έγινε σε μια μεγάλη διάρκεια αλλά σε ένα σχετικά περιορισμένο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό τα αποτελέσματα είναι αξιόλογα, ακόμα πιο αξιόλογα. Ε, όπως σας είπα, τα σχόλια θα τα διαβιβάσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, που ήρθατε εδώ και για την ε, εργασία σας για αυτή τη μελέτη, η οποία θα μας είναι χρήσιμη, παρά τα σχόλια και τις ε, διορθώσεις που σας επισημάναμε για κάποια σφάλματα τα οποία εντοπίζονται στη μελέτη σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για τον κόπο σας και για την παρουσία σας εδώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης και την Επιτροπή Πολιτισμού για την εργασία τους στα τελευταία, τις τελευταίες μέρες. Δεν έχω ανακοινώσεις για τα διάφορα. Θα ήθελα απλώς να σας επισημάνω ότι η επόμενη συνεδρίαση θα είναι την Τετάρτη 25 Απριλίου και στις 25 ε, το πρωί όπου θα έχουμε και ψηφοφορίες. Παρακαλώ φροντίστε όλοι ε, να είναι παρόντα τα μέλη. Σας ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ και τους ε, διερμηνείς για την εξαιρετική τους εργασία, όπως πάντα, και τη Γραμματεία για την καλή προετοιμασία αυτής της ε, συνεδρίασης.